Ευχαριστώ. Okay, colleagues, um, we're Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσουμε τη δημόσια συνεδρίαση. Σα ευχαριστώ που ήσασταν παρόντε στην συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών, αλλά τώρα ανοίγουμε τις πόρτες και περνάμε στη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Θέλω να, χαρα... να χαιρετήσω τον δόκτορα Καρέρα και τον δόκτορα Ραγκάτσι που θα μας παρουσιάσουν τα εθνικά προγράμματα παρακολούθηση στα κράτη-μέλη και την συμβατότητά τους με, τα, με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα δώσω το λόγο στον Σέργιον Καρέρα. Θα ξεκινήσω λοιπόν, αν δεν σας πειράζει. Α, όχι, ο Φραντσέσκο θα ξεκινήσει καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριος Ραγκάτση. Ευχαριστώ και τη γραμματεία της Επιτροπής σας για την πρόσκληση. Η έκθεση αυτή είναι το πόρισμα προκατακτικών ερευνών που έγινε από μια ομάδα ερευνητών το Σεπτέμβριο του 2013. Βασίζεται σε δευτερογενείς πηγές, σε διερευνητική δημοσιογραφία, σε συναντήσεις και συνεντεύξεις με εμπειρογνώμονες για την ψηφιακή και την κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη. Βασιστήκαμε σε έρευνες σε πέντε κρατημέλη, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Σουηδία και κάτω χώρε. Πρώτα απ' όλα σας κάνω μια επισκόψη των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεύτερον θα αναφέρω τα πέντε κύρια στοιχεία που προκύπτουν από την ερευνά μας. Αυτά είναι τα στοιχεία Α και Β στο σχέδιο των ε, ναι. ε, slides μας και ο Σέργιο θα καλύψει τις νομικές πτυχές και τις προτάσεις σε επίπεδο πολιτικής, τα, στοιχεία CKD. Στην έκθεση βλέπουμε να υπάρχουν δύο είδη συλλογής πληροφοριών. Καταρχήν, η παρακολούθηση από τα καλώδια του διαδικτύου υπάρχουν επομένως ε, στοιχεία παρακολούθησης και αναχέτησης ροής των ε, καλωδίων του διαδικτύου, το GCHQ, το αμερικανικό ε, ο αγγλικός φορέας παρακολούθησης υποτίθεται ότι έχει θέσει 200 τέτοιους διακόπτες για την συλλογή πληροφοριών στα καλώδια που πηγαίνουν με τις ΗΠΑ στην Αγγλία αλλά και οι Γάλλοι επίσης στο Τζιμπούτι έχουν αντίστοιχες τέτοιες ε, συσκευές. Το BND, το Γερμανικό Υπουργείο, η Γερμανική Υπηρεσία Παρακολούθηση έχει κάνει το ίδιο και η ΦΡΑ, η Σουηδική Υπηρεσία, κάνει το ίδιο με τα υποθαλάσσια καλώδια μεταξύ Σκανδιναβίας και Ρωσίας. Είναι πρακτικές λοιπόν που είναι παρόμοιες με το πρόγραμμα PRISM στις Ηνωμένες Πολιτείες και οδηγούν στη συλλογή στοιχείων για τους καταναλωτές με τον υποχρεώνται ιδιωτικές εταιρείες που συλλέγουν πάρα πολλά στοιχεία για εμπορικούς στόχους Skype, Google, Facebook κτλ. να δώσουν τα στοιχεία αυτά στις εθνικές αρχές. Ξέρουμε ότι πολλές ευρωπαϊκές υπηρεσίες έχουν ή καταγγέλλεται ότι έχουν αποκτήσει πολλά τέτοια στοιχεία για τους πολίτες τους μέσω αυτού του διάβλου. Όλες οι υπηρεσίες πληροφοριών δεν είναι ίδιες, υπάρχουν διαφορές σε σχέση με τα μέσα που έχουν οι αρμόδιοι πράκτορες στη διάθεσή τους. Αν δούμε λοιπόν τον προϋπολογισμό, αμέσως βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλο πλεονέκτημα της NSA σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς φορείς, πάνω από 7 δισεκατομμύρια εκατομμύρια το χρόνο είναι ο προπολογισμό τους. Στην Ευρώπη η αγγλική υπηρεσία, το GCHQ, είναι περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ που διπλασιάζει τον προπολογισμό άλλων φορέων όπως είναι το BND ή η ΦΡΑ και το ίδιο αν δούμε την απασχόληση. Πόσους εργαζόμενους έχουν αυτοί οι φορείς, δεν υπάρχουν επίσημοι αριθμοί. Υπολογίζεται ότι η ΕΝΕΣ έχει περίπου 37.000 ε, εργαζόμενους χωρίς τους υπεργολάβους, πάνω από 5.600 στο GCHQ και γύρω στις 500 σε άλλους φορείς. Θα τονίσω τώρα πέντε κύριες πτυχές σε σχέση με αυτήν την ε, παρακολούθηση που φάνηκε από την έρευνά μας. Πρώτα απ' όλα Πρέπει να τονίσω ότι η κλίμακα και η διάσταση των προγραμμάτων που έχουν αποκαλυφθεί είναι με άνευ προηγούμενο. Είναι κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές σε ό,τι αφορά τον όγκο των στοιχείων που συλλέγονται και τους τρόπους με τους οποίους γίνεται αυτή η συλλογή και τα είδη στοιχείων που συλλέγονται. Μπορώ να επανέλθω και στην ε, διάκριση μεταξύ δεδομένων και μεταδεδομένων. Τα στοιχεία λοιπόν που συλλέγει μονάχα το GCHQ είναι 21 petabytes την ημέρα. 10 στην 15. Αυτό είναι η ίδια χρήση δεδομένων όπως 2 εκατομμύρια καταναλωτών στο ίντερνετ που χρησιμοποιούν πολύ ε, το διαδικτύο. Ο αριθμός λοιπόν των ατόμων που παρακολουθούνται είναι πάρα πολύ μεγάλος. Ένα δεύτερο σημαντικό θέμα το οποίο δεν γνωρίζουμε πολλά για αυτό το θέμα και αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα σε τεχνικό επίπεδο αλλά και σε νομικό επίπεδο <clears throat> είναι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα συλλεγόμενα δεδομένα και <clears throat> διαβιβάζονται σε τρίτους. Εδώ υπάρχει λοιπόν η διάκριση μεταξύ νόμιμης και παράνομος μορφής παρακολούθησης. Η διάκριση λοιπόν μεταξύ των δύο είναι ασαφής. Γιατί δεν μπορούμε να καθορίσουμε αν αυτά τα οποία γίνονται είναι στοχευμένη ε, παρακολούθηση που είναι απαραίτητη για την αντιτρομοκρατική δραστηριότητα, για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος κτλ. από τη μία πλευρά ή αν είναι χίδιν παρακολούθηση που χρησιμοποιεί τεχνικές data mining, το οποίο παραβιάζει βασικές αρχές ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπάρχουν πολλές κατηγορίες ατόμων που θεωρούνται εκ των προτέρων ύποπτοι και βρίσκονται σε καταλόγους επί τη βάση ερευνών με λέξεις κλειδιά. Τι γίνεται τώρα όταν κάποιος χρησιμοποιεί αυτές τις λέξεις κλειδιά. Επανερχόμαστε στο πρόγραμμα των ΗΠΑ για τη συνολική συνειδητοποίηση σε σχέση με τις πληροφορίες που είχε ε, απορριφθεί από το Αμερικανικό Κογκρέσο το 2003 και 2004. Τρίτο στοιχείο, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό σαν ένα πρόβλημα Ηνωμένων Πολιτειών έναντι Ευρώπης. Τα προγράμματα συλλογής ε, πληροφοριών γίνονται και με συνεργασία μεταξύ συλλεκτικών αρχών Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι λοιπόν μια συντεχνία, ένα συνάφι επαγγελματιών στον τομέα της συλλογής πληροφοριών που συνεργάζονται για τα θέματα αυτά και έχουμε λοιπόν δίκτυα τα οποία βασίζονται σε συμμαχίες μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών. Υπάρχει πολύ στενή σχέση μεταξύ του Βρετανικού και του Αμερικανικού συστήματος συλλογής πληροφοριών, η οποία φάνηκε και από διάφορες ε, ειδήσει στα μέσα ενημέρωσης. Το κύριο ερώτημα εδώ είναι όχι τόσο οι διπλωματικές συζητήσεις μεταξύ των ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θέματα κυρία, εθνικής κυριαρχίας, αλλά για το πώς αυτά τα υπερεθνικά δίκτυα μπορούν να ελέγχονται από αρχές επισκόψεις που να λειτουργούν σε υπερεθνικό επίπεδο. Τέταρτον, αυτά που ξέρουμε για προγράμματα όπως το PRISM είναι ότι δεν είναι μόνο θέματα εθνικής ασφαλείας τα οποία εμπίπτουν, αλλά περιλαμβάνουν και θέματα που έχουν να κάνουν με ιδιωτικές εταιρείες με εταιρικές σχέσεις είτε θεληματικές είτε με το ζόρι. Όταν λοιπόν αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε ως θέματα υβριδικής παρακολούθησης που περιλαμβάνουν και θέματα ασφαλείας αλλά και θέματα εμπορικού συμφέροντος. Αυτά είναι απαραίτητα όχι μόνο για να καταλάβουμε πώς γίνεται αυτή η μορφή παρακολούθησης εμπλέκοντας κανονικούς πολίτες που χρησιμοποιούν το Gmail, το Skype ή το Facebook αλλά επειδή τα θέματα αυτά δεν βρίσκονται στην αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία είναι μέσα στην αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου, θέματα προσωπικών δεδομένων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία εμπλέκονται κατά ανάγκη σε αυτά τα θέματα. Το πέμπτο ερώτημα είναι ότι υπάρχουν τεράστια ερωτηματικά σε σχέση με την λειτουργία μιας ελεύθερης οικονομίας της αγοράς και της δημοκρατικής κοινωνίας. Συλλέγονται πάρα πολλά στοιχεία σε τεράστια κλίμακα, δεν ξέρουμε γιατί επεξεργάζονται από ποιου και προ το όφελο πιανού και με ποιον διαμοιράζονται. Δεν έχουμε καμία εξασφάλιση ότι γίνεται μεγάλη κλίμακα διαδικασία ανάλυση, δηλαδή data mining. Λένε οι υπηρεσίε πληροφορία ότι αυτό είναι για να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία, αλλά ένα κίνδυνο 1% που εμπλέκει 1% των πολιτών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δικαιολογήσει το σπιουνάρισμα των υπολείπων 99% των πολιτών μας. Τα αποτελέσματα φαίνεται ότι είναι Ισχνά, και ακόμα και ο διευθυντής της NSA αναγκάστηκε να πει στο Αμερικανικό Κογκρέσο ότι μόνο μία ή δύο συνωμοσίε διαλευκάνθηκαν και εμποδίστηκαν χάρη στην παρακολούθηση της NSA. Δεν είναι μονάχα λοιπόν αντιτρομοκρατία, υπάρχει και βιομηχανική και εμπορική κατασκοπία η οποία λαμβάνει χώρα και η αναλογικότητα και ο στόχος αυτών των ενεργειών παρακολούθησης είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει. Δεύτερον, τα προγράμματα αυτά υπονομεύουν την βασική εμπιστοσύνη που είναι, τη η βάση της οικονομίας της αγοράς. Είναι και βασικό στοιχείο της δημοκρατικής ζωής και αυτή η δημοκρατική ζωή, η κοινή δημοκρατική ζωή υπονομεύεται αν θεωρούμε ότι όλοι είναι δυνητικά ύποπτοι ο κάθε παίκτη στον οικονομικό χώρο βασίζεται σε μια έννοια εμπιστοσύνη. Αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ επιχειρηματιών και καταναλωτών, ούτε και αυτό μπορεί να αφήσει να λειτουργεί η οικονομία. Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν πλήττονται από αυτές τις ενέργειες. Η ικανότητα των δημοκρατικών καθιστώτων, όπως έδειξε και η Επιτροπή της ΗΠΑ το 1995, βασίζεται στο ότι πρέπει να είναι ισχυρή η διασταυρούμενη έλεγχη. Έτσι διαχωρίζονται τα δημοκρατικά καθεστώτα από τα αστυνομικά κράτη. Οπότε δεν τίθεται μονάχα το θέμα ισορροπίας μεταξύ προστασίας δεδομένων και εθνικής ασφάλειας ή το, στο τεχνικό ερώτημα σε τεχνικά ερωτήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν από εμπειρογνώμονες, αλλά πρέπει να αντιμετωπιστεί και στα πλαίσια του, της φύσης του καθεστώτος και των δημοκρατικών ελευθεριών. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Καρέρα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τα θέματα αυτά. Thank you and, good morning to... Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκλησή σας. Γιατί μας δίνετε την ευκαιρία να σας αναφέρουμε τα συμπεράσματά μας. Νομικές αντιμετωπίσεις. Όλοι γνωρίζουμε τις δικαιολογίες που έχουν βρεθεί για την από τις αστυνομικές και ιδιοκτικές αρχές που λένε ότι πρόκειται για θέματα εθνικής ασφάλειας και δεν έχει καμία σχέση με αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ισχύει όμως αυτό. Ισχύει. η μελέτη μας εξετάζει το κατά πόσον μπορεί να υπάρξει ένας ισχυρότερος, στεναρότερος ρόλος της Ένωσης εδώ και αν είναι απλώς θέμα μόνο των εθνοκρατών μελών. Εμείς προτείνουμε τρεις άξονες. Πρώτον, αναθεώρηση της έννοιας της εθνικής ασφάλειας και της δημοκρατικής νομιμότητας. Όπως έλεγε προηγουμένως και ο συνάδελφός μου. Εδώ πρόκειται για τις αρχές της δημοκρατικής νομιμότητας. Και θα μπορούσαμε να βασιστούμε σε αυτό για να καταλάβουμε τι είναι η εθνική ασφάλεια, τι είναι. Είναι η Ένα από τα βασικά συμπεράσματά μας είναι ότι τα προγράμματα επιτήρηση των κρατών μελών δεν συμβιβάζονται με τη δημοκρατική νομιμότητα και τις αξίες στις οποίες βασίζεται η συνθήκη η εθνική ασφάλεια δεν είναι έννοια που μπορεί πλέον να κατανοείται μόνον από τις κατασκοπευτικές αρχές. Δεν τους ανήκει. Η εθνική ασφάλεια μας επαναφέρει σε εθνικά συντάγματα που είναι βέβαια η βάση της φιλελεύθερης δημοκρατίας των κρατών της Ένωσης και βασίζονται στο διαχωρισμό των εξουσιών. Πρέπει να υπάρχουν λοιπόν έλεγχη και δημοκρατική, δημοκρατική έλεγχη για να δούμε τι κάνουν και τι δεν κάνουν οι αρμόδιες αρχές. Αυτό είναι βασικό για να μην υπάρχουν καταχρήσεις. Εδώ βλέπουμε τα όρια που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα ευρωπαϊκά, στο Ευρωπαϊκό Νομικό Σύστημα που διαχωρίζουν τι είναι νόμιμο και τι είναι παράνομο ως παρέμβαση των κατασκοπευτικών αρχών ή του εκτελεστικού. Και εδώ το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει υπάρξει πολύ δραστήριο και μας έχει φωτίσει για να δούμε τι κριτήρια ισχύουν. Υπάρχει εδώ σοβαρή νομολογία που καθορίζει τα κριτήρια που ορίζουν τι είναι αποδεκτό και τι δεν είναι, τι συμφωνεί με τον νόμο, τι απαιτεί μια δημοκρατική κοινωνία. Υπάρχουν κριτήρια που υπάρχουν σε οποιοδήποτε εκτελεστική αρχή στην Ένωση αλλά και κατασκοπευτική αρχή. Και ως προς το άρθρο 8 λοιπόν της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το άρθρο 5 για τις δημόσιες ελευθερίες είναι πράγματα που δεν πρέπει να τα ξεχνάμε ως προς τις δραστηριότητες των κατασκοπευτικών αρχών. Η Χάρτα των Θεμελιωδών στο άρθρο 51 της αναφέρεται συχνά σαν δικαιολόγηση για αδράνεια, ενώ εφαρμόζεται μόνο στα πλαίσια του ενωσιακού νόμου και εδώ δεν πρόκειται γι' αυτό. Πρέπει να το ξανασκεφτούμε πιο σοβαρά. Η μελέτη αυτή λοιπόν δείχνει ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου έχει θεωρήσει μεν ότι μόνο στα πλαίσια του ενωσιακού νόμου ισχύει η χάρτα, αλλά ότι επειδή βασίζεται και στην παγκόσμια διακήρυξη δεν περιορίζεται σε αυτό. Οι εθνικοί δικαστέ ήδη χρησιμοποιούν τη χάρτα και εκτός των ορίων του ενωσιακού νόμου για να ερμηνεύσουν και να αναθεωρήσουν τις δραστηριότητες, να ελέγξουν τις δραστηριότητες των κυβερνήσεων. Από τον Ιούνιο του 2013 με την Επίτροπο Ρέντινγκ είχαν τεθεί ορισμένα θέματα ως προς την δικαιοδοσία που έχει ένας που δεν έχει καμία δηλαδή νομική δικαιοδοσία. Βέβαια η συλλογή πληροφοριών ή η κατασκοπία και αντικατασκοπία παραμένει εθνικό θέμα, αλλά πρέπει να γίνονται σεβαστές οι ενωσιακές αρχές. Για ποια νου την ασφάλεια μιλάμε, ποια νου. Ο συνάδελφός μου ανέφερε την εμπιστοσύνη, αλλά εδώ δεν πρόκειται μόνο για εμπιστοσύνη, αλλά και για συνεργασία, που είναι και αυτή η βασική αρχή των συνθήκων. Υπάρχουν μέθοδοι συνεργασίες που έχουν παρακαμφθεί επίτηδες. Από το 2003 έχουν συναυθεί πολλές συμφωνίες και όλοι ξέρουμε ότι έχουν υπονομευθεί πολλές συμβατικές υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει. Υπάρχει το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και η παράκαμψη αυτών των αρχών και διάβλων ε, είναι κάτι που υπονομεύει και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο συμπέρασμά μας υπονομεύει την εσωτερική ασφάλεια της Ένωσης στο σύνολό της την εσωτερική λεγό ασφάλεια η κλίμακα της ε, επιτήρησης αυτής υπονομεύει όλες τις αρχές της Ένωσης, τις αρχές που αναφέρουμε τόσες φορές, που δεν είναι μόνο αρχές ηθικές αλλά και νομικές. Είναι υποκλοπή δεδομένων του οποίου και ιδιοκτήτης των δεδομένων αυτών είναι το άτομο. Ίσως να μην είναι η κατάσταση όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά μοιάζει. Και πράγματι από τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη έχουν παρακάμψει όλες αυτές τις αρχές κατάφορα. Τώρα, θέματα διάκρισης. Βλέπουμε ότι σε μερικές χώρες μέλη γίνεται διάκριση μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής υποκλοπής. Η μαζική επιτήρηση αυτήν τη διάκριση την ακυρώνει. Δεν μπορούμε πια να διαχωρίσουμε καθαρά τι είναι εσωτερική και την εξωτερική επιτήρηση των επικοινωνιών. Ας πούμε στη συνεργασία μας με τη ΣΥΠΑ ξέρουμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει μαζέψει στοιχεία για πολίτες του. Πώς μπορούμε λοιπόν να εγγυηθούμε ότι το σύστημα που εφαρμόζεται για τη μυστική επιτήρηση των επικοινωνιών ισχύει και διεθνώς αφού δεν υπάρχει πια τέτοια σαφής διάκριση εσωτερικού-εξωτερικού. Η αρχή λοιπόν της προστασίας των δεδομένων του πολίτη έχει παρακαμφθεί και βλέπουμε πολλές φορές ότι χρειάζονται οι αρχές επιτήρησης και εποπτείας να αντιμετωπίσουν το τη σοβαρή πίεση που υφίστανται για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει δεν υπάρχει μόνο θέμα ανεξαρτησίας αλλά και ανθρωπίνων πόρων. Εδώ βλέπετε τις υπηρεσίες, τις εσωτερικές υπηρεσίες της Ένωσης. Έχουμε ένα όργανο που υποτίθεται ότι συλλέγει πληροφορίες ασφαλείας, το Ίντσεν, αλλά σε ποια νομική βάση στηρίζεται. Δεν υπάρχει. Πρέπει λοιπόν να δούμε και αυτό το θέμα. Αν η Ένωση έχει τη δυνατότητα να συλλέγει στοιχεία για την ασφάλεια, γιατί μας σοκάρει τόσο πολύ το ότι δεν αναφέρουμε την νομική βάση, το νομικό υπόβαθρο. Και η Ευρωπόλ επίσης είναι ουσιώδες να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που χειρίζεται η Ευρωπόλη είναι νόμιμες και έρχονται, προέρχονται από αξιόπιστες πηγές. Δεν υπάρχει τρόπος να το επαληθεύσουμε αυτό. Και αυτό είναι ιδιαίτερα προβληματικό ως προς τις τρίτες χώρες. Νομίζουμε ότι εδώ υπάρχει κάποιο έλλειμμα το οποίο είναι σοβαρό να αντιμετωπιστεί. Επίσης, τι είναι αστυνόμευση και τι είναι συλλογή πληροφοριών ασφαλείας. Οι επαγγελματίες που ασχολούνται με αυτά φαίνεται ότι δεν τα ξέρουν πολύ καλά όλα αυτά. Είναι ασαφή τα όρια. Τώρα στις συστάσεις μας προτείνουμε θεωρούμε σοβαρό να καθοριστούν κόκκινες γραμμές ως προς το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει η Ένωση. Πρώτον, έναν επαγγελματικό κώδικα για τη διαχείριση των δεδομένων, έναν μια επαγγελματική χάρτα. Δεν είναι πια θεμητό να λέμε ότι επειδή δεν έχει δικαιοδοσίες η Ένωση δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι κάτι απαράδεκτο πρέπει να υπάρξει ένας κώδικας που να καθορίζει ποια είναι τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος, όχι μόνο θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως του δικαστηρίου, αλλά και άλλα κριτήρια που να διαφοροποιούν το θεμητό από το αθέμητο, το νόμιμο από το παράνομο. Και ένα ευρωπαϊκό cloud ιδιωτικής ζωής, ιδιωτικότητος που πρέπει να έχει δικές του δικαιοδοσίες ως προς το cloud computing. Μπορεί να μην είναι σφαιρική λύση αυτή, αλλά θα έχει δίνει περισσότερες εγγυήσει προστασίας. Πρέπει δεν να συγχαρούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το σχέδιο κανονισμού του για την προστασία των δεδομένων. Και είναι ζώτικο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να σκεφτεί τις ρήτρε όπως το άρθρο 43 και το 79 ως κόκκινες γαραμές σε διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο. Και μία υποδομή ενωσιακής πολιτικής ώστε να υπάρχει συνεργασία και για τα αντιτρομοκρατικά. Είχαμε ήδη προτείνει ένα σύστημα κυτρίνων καρτών όταν διαπιστώνονται παραβιάσεις που πρέπει να τυχάνουν κάποιας προειδοποίησης. Η συνεργασία πρέπει να χρησιμοποιεί αυτές τις κίτρινες κάρτες και σε περίπτωση επανάληψης κόκκινες κάρτες. ώστε να εφαρμόζονται όντως οι ενουσιακές αρχές και στην προστασία των δεδομένων ακόμη και για τις αντιτρομοκρατικές δραστηριότητες. Και στις συνομιλίες μας με τις ΗΠΑ ίσως να ζητήσουμε τη δημιουργία μιας χάρτας δικαιωμάτων για όλα αυτά τα θέματα. Πρέπει να καταλάβουμε πού υπάρχουν διασυνδέσεις μεταξύ της δραστηριότητας των διοκτικών και αστυνομικών αρχών ώστε να συνεργάζονται πολύ καλύτερα στην ανταλλαγή πληροφοριών. Χρειάζεται περισσότερη υπολογισμότητα εκεί. και λογοδοσία. Ενωσιακή προστασία των whistleblowers και εγγύηση των αιτητών ασύλου. Τον Οκτώβριο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξανασυζήτησε αυτό το θέμα, ζήτησε από την Κομισιόν να αναστείλει τη συμφωνία DFTP. Και νομίζουμε ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του, Υπάρχουν συμφωνίες, σχέσεις εμπιστοσύνης με τις ΣΥΠΑ να αναθεωρηθούν και τα θέματα δικαιωμάτων και ιδιωτικής ζωής να γίνουν προτεραιότητα. Βέβαια Αυτά είναι προκαταρκτικά μόνο. Και από την έρευνά μας πρέπει να μάθουμε περισσότερα, να συνεχίσουμε τις έρευνες, αλλά δυστυχώς οι πόροι που διαθέτουμε είναι αυτοί που αναφέρουμε και στη μελέτη, αλλά πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη, περισσότερη έρευνα για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, τι είδους έλεγχοι εφαρμόζονται, αν εφαρμόζονται από τα κράτη-μέλη Και εδώ ίσως πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τα δεδομένα των κοινωνικών επιστημών. Ευχαριστώ πολύ. Καλά, είναι προκατακτική έρευνα αυτή. Αλλά και μάλιστα σε λίγο χρόνο χρειάστηκε να την κάνουμε. Είναι η δεύτερη μεγάλη μελέτη που είχαμε. Πολύ σφιχτό το χρονοδιάγραμμα. Αν αρχίσετε να το διαβάσετε, συνάδελφοι, θα δείτε ότι οι συστάσεις αυτές είναι, πώς να το πω, είναι αρκετά πολιτικές, έτσι δεν είναι προέρχεται από ένα think tank, μια δεξαμενή νόμιλο προβληματισμού ε, ακαδημαϊκού ε, περιεχομένου, αλλά καλό είναι γιατί αρχίζουμε να σκεφτόμαστε έτσι, κάπως ουσιαστικά για αυτά τα θέματα. Ξέρω ότι δεν είχατε χρόνο να το διαβάσετε οι συνάδελφοι, αλλά θα το διαβάσουν. Δίνομαι στο λόγο στους σκιώδεις ηγητές για να περάσουμε στη συζήτηση που έχουμε μέχρι τις 12 και 4, όπως γνωρίζετε. Άπλετο χρόνο. Ο ήθιστε πρώτα οι σκιώδεις. Ο σκιώδης δηλαδή που βρίσκεται εδώ. Ε, ο Γιάν Άλβρεχτ, ο εναπομείνας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους ομιλητές μας για τη μελέτη αυτή που μας τη παρουσιάσουν σε τόσο επίκαιρο χρόνο. Γνωρίζετε ότι σήμερα ε, γίνεται αντίστοιχη ακρόαση και στη Βουλή των Κοινοτήτων ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, του Διευθυντού της δικής τους υπηρεσίας για να δούμε πώς μπορούμε να τα ελέγξουμε αυτά την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί υπολοιπόμεθα από ό,τι φάνηκε στη συζήτηση την περασμένη εβδομάδα. Και αυτά όλα μας οδηγούν σε κάποιες ευρύτερες και ανώτερες αρχές. Πολύ ξεκάθαρα μας εξηγείται κάποιες συστάσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τι μπορούμε εμείς να κάνουμε, πώς έχει σήμερα η κατάσταση και το εκτιμώ αυτό πάρα πολύ και χαίρομαι. Πραγματικά πρέπει να το μελετήσουμε πάρα πολύ προσεκτικά και να συζητήσουμε εδώ πώς θα αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε και τις συστάσεις αυτές. Δεν θα πρέπει απλώς να παραγωνιστούν και να ξεχαστούν. Και θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν το εξής. Η κατάσταση που έχουμε αυτό το καιρό είναι μια διαρκής παραβίαση των δικαιωμάτων των πολιτών. Τουλάχιστον υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Έτσι, διαρκής, επαναλαμβάνω, παραβίαση των ε, δικαιωμάτων των πολιτών. Και διερωτούμε εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τι μπορούμε να κάνουμε. Ως νομοθέτης δηλαδή συνολικά για να σταματήσει αυτή η παραβίαση και αυτό το περιβάλλον. Διαβάζω ότι στη μελέτη σας εξηγείται βεβαίω και βάσει των αρμοδιοτήτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των εξουσιών τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούν να κάνουν οι αρχέ, συνεργασία αστυνομική με μυστικέ υπηρεσίε, όλα αυτά καλά. Αλλά το ερώτημα που τίθεται είναι πού θα μπουν στη οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Χρειάζονται αλλαγέ εκεί μετά από τις αποκαλύψεις αυτές. Και στη διοργανική γενικότερα εδώ διελκυστίδα που είναι πολιτική υπόθεση θα ήθελα να σας ακούσω να μας λέτε αν ε, τα κράτη-μέλη είναι αρμόδια για κάποιες αρμοδιότητες που δεν έχουμε εμείς. Είχαμε προηγουμένως το διευθυντή της Ίνσεν. Και αυτή η συνεργασία λοιπόν με το κέντρο πώς μπορεί να διαμορφωθεί με το Σίτσεν. Θέλω λίγο να μας ενημερώσετε περισσότερο. Ευχαριστώ. Έχουμε χρόνο. Ε, Οπότε μία ερώτηση, μία απάντηση. Δεν θα ομαδοποιήσουμε, ε, θα απαντάμε οι προσκεκλημένοι μας είτε ο καθένας ξεχωριστά, είτε χωρίστε το όπως θέλετε. Και παρακαλώ να είστε ειλικρινείς. Είστε ε, πανεπιστημιακοί εδώ, δεν είναι το ίντσεν, να μας τα πείτε έξω από τα δόντια. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ναι, εγώ έχω ελευθερία, όχι ως πανεπιστημιακός, ως ανεξάρτητος ερευνητής και θα την αξιοποιήσω. Ε, Σας ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή. η μελέτη προτείνει να αναλυφθεί δράση, πώς να τη χαρακτήσω, πολύ επίπεδη. Δυστυχώς δεν υπάρχει μία απλή λύση. Θα πρέπει το θέμα να ειδωθεί από διάφορες σκοπιές και με διάφορες προσεγγίσεις, αλλά η αφετηρία επανέρχεται στο θέμα της εμπιστοσύνης και της ειλικρινούς συνεργασίας. Τι θα πει αυτό. Το γεγονός ότι δεν μπορούμε πλέον να είμαστε βέβαιοι ότι αυτές οι αρχές και ασφαλιστικές δικλίδες γίνονται σεβαστές που ορίζονται και διανόμου και στις διαπραγματεύσεις όχι μόνο ε, στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά κυρίως σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Ξέρουμε ότι η πληροφορία τη χάνει επεξεργασία σε διάφορα επίπεδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, το PNR αυτή, ε, το θέμα των στοιχείων των επιβατών, υπάρχουν ζητήματα για τα λεγόμενα έξυπνα σύνορα. Smart borders με profiling και χρήση βιομετρικών στοιχείων. Επίσης κάποια ζητήματα που ακούσαμε για οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα θεώρηση της Europol. Ε, δηλαδή αυτό έχει επίπτωση σε ε, πολλά θέματα και πολιτικής που έχει αρμοδιότητα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η μελέτη αυτό συνιστά να αξιοποιήσετε και να εκμεταλλευτείτε τη δυνατότητα που έχετε. Ξεκινούμε από την αρχή της δυσπιστίας και της καχυποψίας. Ε, δεν επιτρέπεται αυτό, θα πρέπει να επανέλθει η εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη δεν είναι δεδομένο. Για τα πρότυπα. Είναι πολύ σαφής η μελέτη να δούμε ποια είναι εκείνα τα πρότυπα που έχουν μεγαλύτερη ε, σημασία. Ε, σαφήνεια, ε, ορατότητα, προβολή του εθνικού νόμου. Ποια είναι τα δικήματα που ψάχνουμε. Γιατί γίνεται αυτή η επιτήρηση και η παρακολούθηση. Το είπε και ο Φραντσέσκο. Γιατί τους παρακολουθούν για την τέλεση κάποιου δικήματος. Ποιο είναι αυτό. Και πώς γίνεται ο έλεγχος και με ποιο τρόπο αντιμετωπίζεται αυτό. Ιδιαίτερα ε, όταν ε, νομοθετούμε θα πρέπει να βλέπουμε ποια είναι η ποιότητα του εκάστοτε νόμου. Είναι βασικό κριτήριο αυτό. Ε, για να δικαιολογείται η νομιμότητα της μυστικής παρακολούθησης από υπηρεσίες ασφαλείας. Επίσης, η ευρωπαϊκή εποπτεία υπάρχει. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, στις υποθέσεις Λίπερ Τσιλίου και Κέννεντι κατά Ηνωμένου Βασιλείου ε, θεώρησε ότι παραβιάζουν τα δικαιώματα και αυτό θα πρέπει να απαντηθεί και από τις υπηρεσίες αυτές. Υπάρχει ένα περιθώριο ελιγμών και βεβαίως υπάρχει ευρωπαϊκή εποπτεία απέναντι σε ε, μια πλήρη ασυδοσία και αυθαιρεσία. Να υπάρχει έλεγχος και από τους εθνικούς, το φυσικό δικαστή. Και επίσης η παρακολούθηση των πολιτών είπαμε ότι δεν έχει να κάνει με την ε, ασφάλεια απέναντι στον ιδιωτικό βίο. Δεν μπαίνει έτσι το δίλημα. Είναι θέμα δημοκρατίας. Θα πρέπει να προστατεύονται οι πολίτες από την αδιάκριτη αυτή παρακολούθηση. Και το δικαστήριο ε, έχει εκδώσει νομολογία έτσι αποφάσει ότι ας πούμε ότι το ανεχόμαστε όταν είναι απολύτως απαραίτητο για τη διαφύλαξη των δημοκρατικών θεσμών. Ισχύει τώρα κάτι τέτοιο. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, να σκεφτούμε ένα κώδικα που θα μπορούσε να εγκρίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Ένωση και να εφαρμόζεται για να προωθείται σε εθνικό επίπεδο. Τώρα, ε, τι γίνεται με την εποπτεία των ε, κρατικών μυστικών υπηρεσιών. Εντάξει, είμαστε ασφαλεί δεν τρέχει τίποτα. Ε, τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο δίκτυο, ε, να εποπτεύουν το ρόλο των μυστικών υπηρεσιών. Υπήρξε και μια δήλωση των Βρυξελών, θυμάστε. Τι απέγινε. Ε, έφερε κανένα αποτέλεσμα. Είναι πιο αποτελεσματική η χρήση της γνώσης και της πραγματογνωμοσύνης που υπάρχει στα εθνικά κοινοβούλια για να ελέγχουν τις υπηρεσίες. Μοιράζονται τις καλές πρακτικές, οι ε, ιδέες τους για να υπάρχει καλύτερη εποπτεία. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος να ε, διαδοθεί ένας τέτοιος κώδικας και να εφαρμόζεται καλύτερα. Η Vivian Redding πρότεινε να υπάρξει μια ευρωπαϊκή υπηρεσία ε, πληροφοριών θα είναι λύση αυτή. Ε, δεν νομίζω. Μια ευρωπαϊκή NSA δεν νομίζω να προσφέρεται για να απαντήσει ε, σε αυτά τα διλήμματα. Η μελέτη όμως λέγει ότι δεν μπορούμε να λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παρακολουθεί. Παρακολουθεί. Βλέπουμε πόσο ανετικές είναι οι επιπτώσεις ε, των όσων συμβαίνουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να προσποιούμαστε ότι δεν τρέχει τίποτα. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα επιχείρημα για να υπάρξει πιο ενισχυμένη και συντονισμένη κοινοτική ένωση, ε, δράση. Και άλλοι συνάδελφοι έχουν ε, τέτοια ερωτήματα. Ο... Η Κάρμεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, νομίζω ότι θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί μιλήσατε με ειλικρίνεια και ελευθερία. Θα προτείνετε στην κυρία Ρέντινγκ να καταγγείλει συμφωνία δικαστικής αρρωγής που δεν έχει οδηγήσει σε τίποτα. Έχουμε μία συμφωνία και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχαμε και τον έλεγχο της συμφωνίας για το TFTP. Θα μπορούσε τώρα η Κομισιόν να κάνει κάτι, να υπάρξει μια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τα θέματα αυτά που θα κωδικοποιήσει καλύτερα αυτές τις συμφωνίες και τι θα κάνουμε με αυτή τη συμφωνία δικαστικής αρρωγής η οποία δεν έχει βοηθήσει σε τίποτα. Θα μπορούσε αυτό να είναι ένα πρώτο βήμα, μια τέτοια καταγγελία για να δείξουμε ποια διαφορά υπάρχει ότι έχουν μια τελείως διαφορετική αντίληψη για τη διάκριση των εξουσιών, για το ρόλο της δικαιοσύνης, για το ρόλο του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω επίσης, δεδομένου ότι μιλήσατε για ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ καυτό σε σχέση με την ιδιοκτησία των δεδομένων. Είναι πράγματι τα στοιχεία αυτά η ιδιοκτησία του κάθε ατόμου, γιατί υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και θεωρίες. Τη στιγμή που δίδει τα δεδομένα αυτά σε κάποιο τρίτο πάβουν να είναι ιδιοκτησία αυτού του ατόμου. Ποια είναι η νομολογία σχετικά με τα θέματα αυτά. Και επίσης κάτι που είναι πολύ σημαντικό σε σχέση με την έρευνά σας είναι το ότι διαλύεται την ε, σύγχυση που υπήρξε μεταξύ των δημοσίων αρχών και των ιδιωτικών αρχών σε ό,τι αφορά την ε, χρήση των δεδομένων αυτών. Φαίνεται ότι εδώ μεγάλο, πρέπει να παίξει μεγάλο ρόλο ο δικαστικός έλεγχος εμείς έχουμε ήδη εγκρίνει μια οδηγία για την προστασία των δεδομένων που δίδει τεράστιο περιθώριο στα κράτη-μέλη. Έχουν μια διακριτική ευχέρεια η οποία είναι τεράστια. Ελπίζω λοιπόν ότι μακάρι να υπήρχε κάποιος κώδικας συμπεριφοράς που να λέει ότι αυτά περιλαμβάνονται μονάχα για ένα, για ένα άτομο το οποίο είναι ύποπτο για κάποιο αδίκημα και όχι γιατί με τον τρόπο αυτό θα συλλέγονται δεδομένα τα οποία θα πολλούνται στις ιδιωτικές εταιρείε. Μιλάμε τώρα για δύο διαφορετικά επίπεδα. Ένα είναι το εμπορικό, ε, η εμπορική κατασκοπία και άλλο είναι η κατασκοπία που ασκείται από τα κράτη-μέλη. Τα ευρωπαϊκά συντάγματα προασπίζουν τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών τους. για να υπάρξει παρακολούθηση στη χώρα μου χρειάζεται δικαστική άδεια. Αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα όμως είναι κάτι το οποίο υπερβαίνει τα εσκαμένα. Δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη τι σημαίνει το Ευρωπαϊκό Σύν, τα συντάγματα των ευρωπαϊκών χωρών. Τα συντάγματα μας έχουν πάψει να έχουν νόημα πια. Είναι μια τεράστια αλλαγή νοοτροπίας που παρακολουθούμε να επισυμβαίνει. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε μια σαφή διάκριση μεταξύ της δημόσιας χρήσης των δεδομένων από τις δημόσιες αρχές για συγκεκριμένους λόγους και η χρήση των ε, ίδιων αυτών δεδομένων από επιχειρήσεις <coughs> και η λειτουργία αυτή συστημάτων όπως αυτό της NSA που συλλέγει και στοιχεία από τις ιδιωτικές εταιρείες είναι ένα περαιτέρω βήμα. <laughs> Βρισκόμαστε τώρα σε μια μετασνοουδενική εποχή όπου τα δεδομένα είναι τελείως διαφορετικά. Ευχαριστώ Κάρμεν. Θέλετε να απαντήσετε στο θέμα αυτό, στο ερώτημα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ένα από τα στοιχεία που τονίζει η έρευνά μας, μία από τις πτυχές της παρακολούθησης και της υποπτίας των αρχών συλλογής πληροφοριών, Κάτι το οποίο τονίζει ε, η ερευνά μας είναι ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών είναι από τη φύση τους, θεωρούν από τη φύση τους δηλαδή, ότι πρέπει να είναι υπεράνω του νόμου. Εμείς το διαμφισβητούμε αυτό, είναι σαφές για μας ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν δέχεται μια τέτοια αντιμετώπιση. Μία από τις προβληματικές πτυχές της μαζικής αυτής παρακολούθησης που αντιμετωπίζουμε είναι το γεγονός ότι, ότι όπως ελέγχθη προηγουμένως εμπλέκεται και η προσωπική ζωή των ατόμων. Γίνεται το λεγόμενο profiling, η ανάλυση δεδομένων που παρακολουθούν τον τρόπο ζωής των ατόμων και προσπαθούν να κάνουν προβλέψεις για την ενδεχόμενη ε, εγκληματικότητα ή δράση τους. Αυτό φαίνεται ότι η απονομική άποψη είναι πάρα πολύ προβληματικό. Είναι κάτι το οποίο πρέπει λοιπόν να αντιμετωπιστεί και να βρεθεί κάποια λύση για αυτά τα θέματα. Στι ΗΠΑ υπήρξαν συζητήσεις για το συνδυασμό διαφορών ενεργειών ανάλυσης δεδομένων, το αναφέρουμε αυτό στην έκθεσή μας, έχει υπάρξει μια εστίαση στο γεγονός ότι η συλλογή δεδομένων θα πρέπει να αφορά μοναχά άτομα τα οποία υπόκεινται σε έρευνες, είναι υπό έρευνα δικαστικού χαρακτήρα ή άλλου χαρακτήρα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το τονίσουμε η ιδιοκτησία των δεδομένων. Νομίζω ότι ο κανονισμός για τα προσωπικά δεδομένα που έχει εγκριθεί και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ιδιαίτερα στεναρό από αυτή την άποψη και αυτό το χαιρετίζω. Ένα αντίστοιχο καθεστώ. θα πρέπει να εφαρμόσετε και στι δραστηριότητε των διοκτικών αρχών. Φυσικά. Μπορούμε να κάνουμε κι άλλο ένα γύρο και να επανέλθουμε στα θέματα αυτά. Η κυρία Μορβάη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ βάλτε τα ακουστικά σας για να ακούσετε τα ουγγρικά μου. Όταν υπήρξε η δημοκρατική μετάβαση στην Ουγγαρία, είχαμε ένα προσκεκλημένο που ήρθε από τη Δυτική Ευρώπη και μας είπε το εξής. Ο κομμουνισμός είναι ένα σύστημα που είναι σαν μια βραδινή παράσταση. Όλοι παρακολουθούν τι γίνεται, αλλά όλοι ξέρουν ότι είναι απλώς ένα θέατρο, ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι πραγματικότητα. Το ίδιο πράγμα γίνεται και με τις δυτικές δημοκρατίες. Εμείς νομίζαμε τότε ότι υπήρχε ένας άλλος κόσμος έξω από το κομμουνιστικό στρατόπεδο, πέρα από το σιδηρούν παραπέτασμα, ότι εκεί υπήρχε δημοκρατία, κράτος δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα και ότι όλα αυτά τα πράγματα ίσχυαν στη Δύση. Και όλα αυτά είναι απλώς μια παράσταση, είναι απλώς μια θεατρική παράσταση και εδώ στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν έχουμε λοιπόν ένα τόσο σημαντικό θέμα από 120 μέλη της Επιτροπής μας είναι μονάχα 7 ή 8 που είναι παρόντα όταν πρόκειται για ένα τόσο σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με την δημοκρατία. Τώρα που είναι 11 και 4, σας λέω, 8 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι παρόντα. Πού είναι ο κύριος Σταβάρες, Δεν αγωνίζεται για τη δημοκρατία ο κύριος Σταβάρης. Τα άλλα μέλη του, της ομάδας μας δεν ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Ασχολείται όμως με την Ουγγαρία, δεν ασχολείται με την παρακολούθηση των Ευρώπαιων πολιτών. Ίσως οι συστάσεις που θα διατυπώσετε θα μπορούν να περιλαμβάνουν την ανάγκη να εξετάσουμε προσεκτικότερα τις αξίες, την ιδεολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δυτικής Ευρώπης και πώς είναι διαφορετικές από την ε, κομμουνιστική εποχή που ξέραμε τουλάχιστον μας παρακολουθούσαν σε κουριτάτε, στάζι, ξέραμε ότι μας παρακολουθούσαν και ήταν δεδομένο αυτό. Είναι και πάλι σας λέω μόνο οκτώ μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρόντα το λέω αυτό για αυτούς που βρίσκονται στο διαδίκτυο και μας παρακολουθούν. Όταν υπήρχε κομμουνισμός παρακολουθούσαν όλους τους πολίτες με ισοδίκαιο τρόπο και ήταν τμήμα του συστήματος ότι ήταν προφανές ότι υπήρχε μαζική παρακολούθηση των πολιτών. Ακόμα θέλουμε να εξασφαλίσουμε στην Ουγγαρία ότι θα δημοσιευθεί ο κατάλογος των πρακτόρων. Προσπαθούμε να ξαναβρούμε την αλήθεια, να δούμε ποιον είναι το παρελθόν μας, τι έχει γίνει. Ποιοι ήταν οι ένοχοι οι οποίοι παρακολουθούσαν στην κομμουνιστική εποχή όλο τον κόσμο. Και τώρα εδώ στη Δύση λένε όχι δεν παρακολουθείται κανένας, δεν παρακολουθούνται τα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία, ότι δεν υπάρχει μαζική παρακολούθηση. Αλλά είναι τόσο φυσικά όλα αυτά που γίνονται, ώστε οι συνάδελφοί μου δεν αδειάσουν να έρθουν σε μια τέτοια συνεδρίαση. Δεν τους ενδιαφέρει ότι είναι κάτι τέτοιο. Δεν νιώθουν καμία εντύπωση για όλα αυτά. Κάποιος είπε στην προηγούμενη συνεδρίαση ότι όλα αυτά είναι απόλυτα φυσιολογικά και δεν καταλαβαίνει γιατί υπήρξε τόση φασαρία για όλα αυτά. Μήπως θα πρέπει λοιπόν να ψάξουμε περισσότερο στα θέματα αυτά. Δεν υπάρχει πια κάποιο ασφαλές καταφύγιο σε κανένα από τα κράτη-μέλη μας. Ίσως η Ουγγαρία θα πρέπει να δώσει πολιτικό άσυλο στον Σνόουδεν, γιατί μας έδειξε ότι όλα αυτά είναι απλώς μια παράσταση, μια φενάκι. Έφερε τελικά την αλήθεια μπροστά σε όλους μας και μας έδειξε ότι ο βασιλιάς είναι γδιτός, είναι τσίτσιδος. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν τι ακριβώς σημαίνει η δημοκρατία και εσείς ως ακαδημαϊκοί θα πρέπει να προτείνετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ξανασκεφτεί τι είναι η δημοκρατία και πώς λειτουργεί. Ευχαριστώ. Uh, point of order from Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να πω εδώ ξεκάθαρα ότι δεν επιτρέπεται τέτοια συμπεριφορά απέναντι σε συναδέλφους ιδιαίτερα απόντες. Είναι τελείως ανάρμοστο. Ε, θα πρέπει σοβαρά να ασχοληθούμε με το θέμα και όχι με λαϊκιστικές απόπειρες και πυροτεχνήματα να προσπαθούμε να ε, καθιστούμε υπεύθυνου με μονομένους βουλευτές για αυτό που αποφάσισε η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου μου για τη σχέση και την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουγγαρία. Το ξέρω ότι μπορεί να υπάρχει ένα σημείο βουλευτή που να μην είναι ευχαριστημένη με αυτά που λέει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την παραβίαση των θεμελιωτών δικαιωμάτων στην Ουγγαρία και ε, αλλού στην Ένωση. Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, να κάνουμε, αλλά ε, θα πρέπει να συνεννοηθούμε για μια συμπεριφορά που θα έχουμε ένας απέναντι στον άλλον για να συζητούμε ε, σοβαρά και να μην επιτιθέμεθα ένα στον άλλον έτσι με φωνασκίες και άλλα τέτοια. Uh, Καλά, τώρα δεν θέλω να μπω σε τέτοια συζήτηση, αλλά ακριβώς όταν έχουμε από όντα μέλη δεν είναι σωστό να αναφερόμαστε. Και ούτε φταίω που λείπει, λέει η κυρία Μορβάη. <laughs> Εντάξει, το είπατε. Ακούστηκε και η απάντηση, ο λόγο βουλευτής απουσιάζει. Λοιπόν, δεν θέλω να το κάνουμε τώρα θέμα. Ακούστηκαν δύο απόψει και ο ελόγου βουλευτής είναι απόν. Είναι άδικο απέναντί του να το συζητάμε. Αυτά. Ας προχωρήσουμε. Ε, θα απαντηθεί στη συνέχεια αυτό που ρωτήσατε. Ε, ο κύριος Βάιντεν Χόλτσερ. Νομίζω ότι ε, θα ήταν πολύ καλό και θα γνώριζε περισσότερη προσοχή αυτό που μας απασχολεί εδώ ε, εάν υπήρχε ευρύτερη διάδοση. Και χαίρομαι και ευχαριστώ πολύ ε, για την ποιότητα της μελέτης αυτής. Είναι πάρα πολύ συστηματική, αξιόλογη και μας δίνει μεγάλη τροφή για σκέψη και θα έπρεπε να προβληματιστούμε κιόλας. Όλο και περισσότερο έχω εγώ την αίσθηση ότι τώρα βρισκόμαστε στην εξής ιστορική στιγμή και κατάσταση. Δεν πρόκειται μόνο για την ευέλεια αυτού του σκανδάλου, αλλά για πολύ πιο ε, ε, θεμελιώδη θέματα, η ελευθερία των πολιτών, των κρατών και η ελευθερία των καταναλωτών ακόμα. Είναι αυτή που κυβεύεται. Και πραγματικά ε, είναι τεράστιες οι αλλαγές και εξελίξεις και θα πρέπει κανονικά να απασχολήσουν και το Κοινοβούλιο. Κάτι που με ανισχύει ιδιαίτερα και με έχει θορυβήσει είναι αυτή η ανάμειξη και η σύγχυση που γίνεται ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό βίο. Υπήρχε βέβαια και στο παρελθόν όπου κανείς παρακολουθούσε τους ιδιώτες Πολύ ωραία αναφερθήκατε σε αυτή την αναγκαστική συνεργασία, αλλά υπάρχει και μια θελοντική συνεργασία. Και αυτό το δεύτερο στοιχείο είναι κάτι ε, πολύ προβληματικό. Πού είναι εδώ το θελοντικό στοιχείο. Και μάλιστα όταν συνεργάζονται ε, και ο θελός οι εταιρείε επιβραβεύονται. Όχι με χρήμα, γιατί δεν είναι το χρήμα πλέον ε, το νόμισμα ε, σε αυτές τις συναλλαγές στο σύγχρονο κόσμο, αλλά τα δεδομένα. Ε, και αυτό είναι το κέρδος που αποκομίζει μια εταιρεία όταν συνεργάζεται. Θα με ενδιαφέρει λοιπόν να μας λέγατε περισσότερα γι' αυτά. Είπατε ότι δεν γνωρίζετε πολλά πράγματα για αυτή την επεξεργασία των δεδομένων, αυτό το processing και πώς γίνεται αυτή η συλλογή τους. Αλλά κάτι θα έχετε ακουστά. Υπάρχουν κάποιες παρακολουθήσεις που με ενδιαφέρουν και τις έχω ψάξει και δείχναν ότι υπάρχουν εταιρείες που ασχολούνται πολύ εντατικά ε, με τη διαχείριση αυτών των δεδομένων, την επεξεργασία τους. Είναι μια εκεί πραγματικά για να κάνει ε, κάποιος διαφήμιση σε συγκεκριμένους ανθρώπους, στοχευμένα, και δεν υπάρχει συμμετρική ας πούμε πληροφόρηση, ενημέρωση, ακόμα και διαφήμιση για την αγορά. Στοχευμένα από την αρχή δεν με θεωρούν πολίτη αλλά καταναλωτή. Και δεν καταργείται έτσι μόνο το αστικό κράτος αλλά και ολόκληρη η οικονομία της αγοράς. Διότι δεν είμαστε πλέον σε θέση να λαμβάνουμε ε, προσωπικές αποφάσεις. Τώρα δεν θέλω να χαθώ σε φιλοσοφικές αναλύσεις, αλλά είναι πραγματικά πολύ συγκλονιστικά όσα συμβαίνουν και η μελέτη εξάλλου πολύ καλή και πρόκειται για την εσωτερική ασφάλεια του συνόλου της Ένωσης. Μα αυτό είναι το θέμα μας ακριβώς. Τα όσα συμβαίνουν τώρα παράγουν ανασφάλεια στον κόσμο. Υποτίθεται ότι μας περισσότερη ασφάλεια, αλλά δημιουργείται ε, τέτοιος όγκος ανασφάλειας που δεν έχει ε, ε, εμφανιστεί ποτέ στο παρελθόν. Είναι άνευ προηγουμένο αυτά το φαινόμενο. Και παρακαλώ αυτό το θέμα της συνεργασίας των δημοσίων, των κρατικών με τις ιδιωτικές εταιρείες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή για να θέσω και εγώ το ερώτημα που ακολουθεί ο κύριος Χίνγκστρομ, αλλά προηγουμένως. κύριε Χίνγκστρομ, ε, θα ήθελα να θέσω και εγώ το ερώτημά μου. Γιατί ο κ. Βάιντερ Χόλτσερ άρχισε να μπαίνει στα θέματα, τα θέματα σχέσεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Πιστεύω και εγώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμη η μελέτη σας και εσείς ε, τονίσατε ότι είναι μια προκατακτική μελέτη. Σε ένα πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έχει εκπονηθεί αυτή η μελέτη. Αλλά θέλω να θέσω αυτό το σημαντικό ερώτημα για τους λεγόμενους ασφαλεί ασφαλείς λιμένες που αντιμετωπίσαμε σε μία από τις ακροάσεις μας και ήταν ιδιαίτερα έντονα αυτά τα οποία ακούσαμε. Και επίσης όλες οι εταιρείες που εμπλέκονται στο πρόγραμμα Prism, Google, Facebook κτλ. είχαν ήδη υπογράψει τη συμφωνία αυτή για τον ασφαλή λιμένα. Ποια είναι η δική σας άποψη τώρα για το θέμα αυτό. Τι μπορεί να διασωθεί από αυτό το, τη συμφωνία του Safe Harbor. Μπορείτε να μιλήσετε και για κάτι αυτά που είπε ο Γιώζεφ. για το ρόλο των παρόχων υπηρεσιών και για τις συνέπειες για, το, για τον εμπορικό χώρο. Εμείς πήγαμε στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή εμπορίου την FTC στις Ηνωμένες Πολιτείες και μιλήσαμε για την έλλειψη, για την κατάρρευση της εμπιστοσύνης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και σε εμπορικό επίπεδο υπάρχει μια τεράστια κατάρρευση εμπιστοσύνης. Στη μελέτη σας βέβαια, εσείς βέβαια δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε το τεράστιο αυτό θέμα της ε, κατάρρευσης των εμπορικών, της εμπιστοσύνης μεταξύ εμπορικών εταίρων. Εσείς όμως έχετε την ακαδημαϊκή ελευθερία, μπορείτε να μας δώσετε μια ευρύτερη εικόνα για το τι συμβαίνει στον τομέα αυτό. Και δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσετε και μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο Εγκ Ευχαριστώ πολύ. Όλα αυτά είναι σημαντικά ερωτήματα τα οποία θέτετε και εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά τα στοιχεία και να σας πω τι ξέρουμε αυτή τη στιγμή και τι δεν ξέρουμε προς το παρόν, τι πρέπει να μάθουμε ακόμα. Κάτι το οποίο ξέρουμε σίγουρα και αυτό συζητήθηκε σε πολλούς ε, επιχειρηματικούς κύκλους και σε τεχνολογικό επίπεδο. Το νέο χρυσάφι, το νέο πετρέλαιο είναι τα δεδομένα για τον αιώνα μας. Μια βασική αρχή λοιπόν θα πρέπει να είναι ότι όλες οι εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούν τα δεδομένα αυτά <clears throat> σαν κύριο στοιχείο του επιχειρηματικού τους μοντέλου όπως είναι το Facebook, το Google και πολλές άλλες εταιρείες οι οποίες δεν είναι τόσο γνωστές, οι οποίες όμως κάνουν μαζική επεξεργασία δεδομένων, παραγματικά τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες. Όλοι αυτοί λοιπόν βασίζουν την εργασία τους στην εμπιστοσύνη. Στην εμπιστοσύνη ότι οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις θα κρατήσουν εμπιστευτικά τα δεδομένα. Οι αποκαλύψεις όμως τώρα έδειξαν ότι αυτό δεν ισχύει. Έχει διαβρωθεί κάθε εμπιστοσύνη που μπορεί να έχει ο καταναλωτής σε σχέση με το πώς τα δεδομένα των καταναλωτών τη χάνουν επεξεργασίες από τις εταιρείες αυτές λόγω της φύσης των σχέσεων που μπορούν να έχουν με ευαγή ιδρύματα όπως η NSA, αλλά όχι μόναχα, με το GCHQ στο Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες υπηρεσίες πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έλεγα λοιπόν ναι και αυτό το τονίζουμε στη μελέτη μας διακυβεύονται οι ατομικές ελευθερίες, διακυβεύονται τα δικαιώματα των καταναλωτών και αν το δούμε από την οπτική γωνία των επιχειρήσεων τίθεται να αμφιβόλω η οικονομική βιωσιμότητα των εταιριών. Και αυτό μπορεί να μην είναι το πιο σημαντικό, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αναφέρουμε. Ότι οι πρόσφατες δηλώσεις του επικεφαλής της Google σε σχέση με τα θέματα αυτά είναι εύγλωτες. Γιατί φαίνεται ότι η NSA όχι μόνο θα τους υποχρεώσει εταιρείε όπως η Google να δίδουν συνέχεια στις αιτήσεις τους, αλλά ότι επίσης έχουν παρακολουθήσει και στοιχεία μεταξύ διαφορετικών διακομιστών της Google που δεν ήταν κωδικοποιημένα γιατί θεωρείται ότι ήταν μια ασφαλή σύνδεση και αυτό δεν έχει γίνει μόνο στις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν μιλάμε για μετάδοση δεδομένων μεταξύ διαφορετικών κέντρων δεδομένων της Google μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου υπήρξε παρέμβαση της NSA. Και η απάντηση του επικεφαλής Google ήταν αγανάκτηση γιατί εδώ εμπλέκονται σημαντικά εμπορικά συμφέροντα. Για να ξαναγυρίσω τώρα στη σχέση μεταξύ εταιριών και υπηρεσιών πληροφορίας, πληροφοριών, θέτεται σημαντικά ερωτήματα για τα οποία εμεί όμως δεν έχουμε τις απαντήσεις προς το παρόν και αυτό θα απαιτήσει πολύ περισσότερη έρευνα βέβαια. Αυτό που ξέρουμε είναι το πρόγραμμα PRISM των Ηνωμένων Πολιτειών και πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι τα δεδομένα αυτά είναι διαθέσιμα και στην Αγγλική Υπηρεσία Πληροφοριών μέσα στην, στο πλαίσιο της συμφωνίας που έχει το GCHQ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, τη λεγόμενη πενταματική συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων, Ηνωμένων Βασιλείου, Νέας Ζηλανδίας, Αυστραλίας και Καναδά. Πρόκειται λοιπόν για μια υπηρεσία πληροφοριών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι όλα αυτά που γνωρίζει το GCHQ ε, μέσω του προγράμματος PRISM μπορεί να τα γνωρίζουν και άλλες υπηρεσίες πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά τα δεδομένα λοιπόν δυνητικά είναι δεδομένα πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το είδο λοιπόν της ε, εποπτείας που ασκείται από τις υπηρεσίες πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται πράγματι μέσω αυτών των υβριδικών εταιρικών σχέσεων υπηρεσιών πληροφοριών με ιδιωτικές εταιρείες. Να σταθώ τώρα για δύο άλλα σημεία. Για το αν αυτές οι εταιρείε θεληματικά συνεργάζονται ή υποχρεώνται να συνεργάζονται. Έχουμε στοιχεία ότι έχουν υποχρεωθεί με νομικό τρόπο να συνεργάζονται, αλλά δεν ξέρουμε πόσες από αυτές οι εταιρείε έχουν με εθελοντικό τρόπο προτείνει τις υπηρεσίες τους. Υπάρχουν όμως και εταιρείε που έχουν αποφασίσει να αντισταθούν, ίσως όχι πολλές, κάποιες εταιρείε η Levebit, παραδείγματος χάρη, ή το Silent Circle έχουν αρνηθεί να ε, συμμετάσχουν σε αυτά τα προγράμματα. Η Levebit έδινε ε, υπηρεσίες κωδικοποιημένων ε, ηλεκτρονικών ταχυδρομείων και η εταιρεία αυτή αποφάσισε να κλείσει και όχι να υπακούσει σε μια ε, νομική αίτηση για να δώσει δεδομένα και τώρα ο επικεφαλής της κινδυνεύει με νομική δίωξη γιατί δεν έχει συνεργαστεί. Υπάρχει λοιπόν υψηλό κόστος που πληρώνει κανείς αν δεν συνεργάζεται. Και ίσως μπορώ να σταματήσω εδώ και να αφήσω τον Σέρχιο να ανεφερθεί στο θέμα του Safe Harbor. Ο κύριος Έγκστρομ περιμένει με υπομονή να θέσει το ερώτημά του και ίσως μπορείτε να απαντήσετε και στα δύο μαζί κύριε Έγκστρομ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ραγκάτσι, με ενδιέφερε αυτό που είπατε για την χρησιμότητα αυτής της μαζικής παρακολούθησης. Είπατε καταρχήν ότι η NSA είπε ότι για κάπου 54 περιπτώσεις που οδήγησε σε ε, αντιμετώπιση συνωμοσιών τρομοκρατών, αλλά τελικά κατέληξε σε δύο-τρεις μονάχα περιπτώσεις που απέτρεψαν κάποια τρομοκρατική ενέργεια. Φυσικά είναι πολύ σημαντική η τρομοκρατία. Mm. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα. Οι έκτακτες παραδόσεις της CIA αναφέρθηκαν κτλ. Αλλά αν βρεθεί μια πραγματική συνωμοσία τρομοκρατικού χαρακτήρα, θα περίμενα να τους φέρουν στα δικαστήρια και να υπάρξουν κάποιες καταδίκες. Έχουν οδηγήσει αυτές οι περιπτώσεις μία-δύο σε καταδίκες στις ΗΠΑ. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημά μου. Το δεύτερο ερώτημα είναι στη Σουηδία. Η κυβέρνησή μα λέει παρόμοια πράγματα ότι η παρακολούθηση από την FRA έχουν αποτρέψει πολλέ αρνητικέ ενέργειε, αλλά δεν έχουν δώσει καθόλου, καθόλου λεπτομέρειες και δεν έχουν αναφέρει οποιαδήποτε υπόθεση που είναι ενώπιον των Σουηδικών δικαστήριων. Γνωρίζετε εσεί κάποια περίπτωση στα Σουηδικά δικαστήρια όπου υπήρξε δίωξη λόγω αυτών των παρακολουθήσεων. Ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι η NSA μας αποκάλυψε συγκεκριμένες περιπτώσεις, δεν το ξέρουμε. Δεν γνωρίζω δηλαδή ειδικές δικαστικές υποθέσεις. Δεν σημαίνει ότι δεν ισχύουν, απλώς δεν τις ξέρω εγώ. Αλλά αυτό είπαμε και εμείς ότι χρειάζεται περαιτέρω μελέτη για ακριβώς τέτοιου είδους στοιχεία. σύντομα να επανέλθω σε αυτό που είπατε πριν για τη Συμφωνία Ένωσης ΕΠΑ, ΕΕ, Safe Harbor. Η συμφωνία αυτή έχει παραβιαστεί κατάφορα και πρέπει να σκεφτούμε τρόπους να δούμε πώς θα μπορούσε το cloud computing να χρησιμοποιηθεί Να δούμε δηλαδή αν υπάρχουν επαρκείς δοκιμές. Ο κύριος Κρούνεν. Μήπως όμως ξέρετε και καμία περίπτωση προμηθευτών ίντερνετ που να έχουν παραβιάσει τα ισχύοντα η France Telecom ίσως. Καλέσαμε μεγάλους προμηθευτάς όπως τη France Telecom αλλά δεν έχουν έρθει. Μήπως μπορείτε να το σχολιάσετε και αυτό. Κύριε Καρούνα, θέλετε να πείτε τίποτα. Ε, όχι, ήθελα απλώ να σας συγχαρώ ε, για την μελέτη αυτή που μας παρουσιάσατε. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα είναι και θα τη διαβάσω πολύ προσεκτικά. Δεν ξέρω, ίσως η απάντηση της ερώτησής μου να βρίσκεται στην έκθεση αυτή τη μελέτη, αλλά πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγο καιρό ο πρώην καγκελάριος Σρέντερ της Γερμανίας σε μια συνέντευξη που το ρώτησαν ε, ε, τι ε, κάνει και με τι ασχολείται και ε, ποιες είναι οι εργασίες του. Ήξερε απολύτως ότι του παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα και ήξερε ότι ήταν τελείως ε, αδύνατο ε, να ξεφύγει από τις υποκλοπές και το, το φακέλωμα. Λοιπόν, έχω να σας ρωτήσω το εξή: Τι μπορείτε να προτείνετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε να εκπονήσει ένα πρότυπο, έναν κανόνα, μια στρατηγική για να προλαμβάνει τέτοια φαινόμενα. Αυτή τη στιγμή θεωρούμε ε, ότι δεν μπορεί κανείς να ε, εμποδίσει τις υποκλοπές και τις παρακολουθήσεις. Τι μπορούμε να κάνουμε για να αποτρέψουμε ε, κάποιους από τη χρήση τέτοιων πληροφοριών, είτε αυτές είναι εμπορικές χρήσεις είτε άλλες. Εντάξει, υποκλέπτονται, αλλά τουλάχιστον να μην χρησιμοποιούνται μετά. Επίσης συμφωνώ απολύτως όταν λέτε ότι θα πρέπει να αλλάξει αυτή η έννοια της εμπιστοσύνης και να κινούμε από τη δυσπιστία και την καχυποψία. Αυτό είναι το δεδομένο και το ζητούμενο είναι η εμπιστοσύνη. Όλα αυτά τα χρόνια εμείς πιστεύαμε ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας ήταν η προτεραιότητα, είχαμε εμπιστοσύνη και μάλιστα υπερβολική θα έλεγα μέχρι και αφέλεια επιδείξει για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Και πολλοί υπερέβαλαν και ξεπέρασαν και τα αιτήματα των διαφόρων ε, ε, υπηρεσιών ασφαλείας, πληροφοριών και των κρατών ακόμα. Um, first... Λοιπόν, Μήπως να απαντήσω πρώτα σε αυτό και θα επανέλθω στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση αυτή. Είναι πολύ σημαντική. Γιατί και οι ιδιώτες ε, διαρωτώνται πώς μπορούν να προστατεύσουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Υπάρχουν τεχνικοί τρόποι σε επίπεδο ατόμου φυσικά, φυσικού προσώπου. Δηλαδή, το δίκτυο TOR είναι καλό για να προστατεύσεις το προσωπικό σου διαδίκτυο από την κατασκοπία. Υπάρχουν τεχνολογίες που δεν έχει καταφέρει η NSA συστηματικά να σπάει. Υπάρχουν και λογισμικά ανοιχτής πηγής, δωρεάν δηλαδή, ε, ε, κρυπτογράφησης και δεν κατάφερε ούτε αυτά η NSA να τα σπάσει ακόμα. Παρόλο που έχουν αφιερώσει ε, σημαντικά ποσά. Για να μπουν ε, από διάφορα παραθυράκια σε συστήματα ιδιωτικά για κρυπτογράφηση. Διάβασα στο blog του υπαλλήλου της Google ε, που δήλωνε ότι για το Gmail, για τη διεύθυνση ε, το email των ιδιωτών χρειάστηκε δύο-τρία χρόνια ε, για να μπορέσει να εξασφαλίσει ότι παραμένουν ασφαλή και με κρυπτογράφηση. Υπάρχουν λογισμικά λοιπόν open source που μπορούν να εξασφαλίσουν ένα στοιχειώδες επίπεδο ιδιωτικού βίου. Σε πιο ε, διαρθρωτικό επίπεδο τώρα είναι να δημιουργηθεί ένα cloud στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ιδιωτική ζωή που δεν εξασφαλίζει 100% ιδιωτική ζωή αλλά μπορεί να φέρει περισσότερη προστασία στα προσωπικά δεδομένα ε, των πολιτών. Υπάρχουν και τεχνικές αντίστοιχες. Δηλαδή, ε, αποθηκεύεις σε ένα cloud τα δεδομένα σου και τα στέλνεις κάπου χωρίς να περνάνε απαραίτητο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν άλλα δίκτυα και άλλες τεχνικές λύσεις ε, που προτείνουμε στη μελέτη. Για να απαντήσω σύντομα και κάτι ε, περισσότερο από την τεχνολογική πλευρά, ο συνάδελφος θα απαντήσει τα νομικά. Ο Βίλιαμ Μπίνι, ε, whistleblower της NSA, ε, καταγγέλων, εξήγησε ότι το 2000 υπήρχε μια τεχνολογία που είχαν αναπτύξει αυτός και συνάδελφοί του έτσι ώστε πάνω κάτω να κάνουν αντίστοιχα με αυτά που γίνονται τώρα ως προς την παρακολούθηση και τη δυνατότητα ανείχνευσης ε, των ιχνών που αφήνουν οι πολίτες στο διαδίκτυο χωρίς μαζική αποθήκευση δεδομένων, χωρίς αυτό το μαζικό φακέλωμα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Υπήρχε λοιπόν ένα τέτοιο πρόγραμμα ε, που ε, είχε το Privacy by Design. Το απέριψε αυτό η NSA <laughs> και μας ε, είπε ότι προφασίστηκαν οικονομικούς λόγους. Όταν έχεις ένα τεράστιο πρόγραμμα που να αποθηκεύει εκατομμύρια δεδομένα θα χρειαζόταν ε, τεράστιους προϋπολογισμούς και αυτό χρειαζόταν τότε η NSA. Λοιπόν, δεν λέω απολύτω εγώ κατά ανάγκη ότι δεν θα πρέπει να εμπιστευόμαστε τι μυστικέ υπηρεσίε στην καταπολέμηση τη τρομοκρατία ή όταν λένε ότι είναι προτεραιότητά του. Είναι. Ε, ε, προφανώς, αλλά υπάρχει και ένα θέμα αναλογικότητας και ο στόχος, για ποιο σκοπό συλλέγονται όλα αυτά τα στοιχεία, θα πρέπει κάπου να συμβαδίζουν οι εξέλιξεις, διότι οι τεχνολογίες έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν και μπορείς να επιτύχεις τον ίδιο στόχο χωρίς όλη αυτή την άχρηστη συλλογή όλων αυτών των ιδιωτικών δεδομένων και στοιχείων των πολιτών. Μια τελευταία ερώτηση ε, της κυρίας Σίπελ και συμπληρωματική του κύριου Άλμπρεχτ. Σας ευχαριστώ. Να ξαναγυρίσω στο ερώτημα για την ε, διεύρυνση της συλλογή δεδομένων. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν μέχρι στιγμή στοιχείο της ερευνάς σας για μένα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξετάσουμε περισσότερο τη διάσταση της ε, παρακολούθηση και αν αυξήθηκε αυτή η διάσταση μετά τις επιθέσεις της 11 ε, Σεπτεμβρίου και επίσης ακόμα και αν εξακολουθεί να υπάρχει και υπήρχε και πριν αυτή η παρακολούθηση αν πράγματι είναι ανάλογη, αν υπάρχει αναλογικότητα με το αποτέλεσμα που έχει επιτευχθεί σε ό,τι αφορά την ε, αποτροπή ε, απαντήσεων, τρομοκρατικών ενεργειών. Και έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο προπολογισμό τη NSA και έχει πράγματι αποτραπεί τόσο πολύ η τρομοκρατία ή έχει γίνει τόσο πολύ πιο ασφαλή η ζωή στι ΗΠΑ λόγω τη χρηματοδότηση αυτή τη NSA. Θα ήθελα λοιπόν να απαντήσετε για τα θέματα αυτά. Και <clears throat> χαίρομαι για αυτό που είπατε ότι σίγουρα πρέπει να υπάρξει μια ευρωπαϊκή αρμοδιότητα για τη λειτουργία των μυστικών υπηρεσιών, αντιμετωπίσουμε πάντα το ερώτημα τι νόημα έχουν οι νόμοι μας και οι κανόνες μας αν είναι μια υποψία τεκμηριωμένη ότι κάποιες μυστικές υπηρεσίες δεν τηρούν κανένα από αυτούς τους νόμους. Λοιπόν, όταν υπάρχει υποψία ότι κάποιοι δεν τηρούν ποτέ φλήρως αυτούς τους νόμους, τι νόημα έχει να νομοθετούμε. Γι' αυτό είναι ενδιαφέρουσες οι κόκκινες γραμμές που έχετε αναφέρει σε σχέση με το ρόλο των μυστικών υπηρεσιών και το ερώτημα το οποίο, <clears throat> δεν, το οποίο τίθεται δεν είναι μονάχα το θέμα του να έχουμε κόκκινες γραμμές αλλά πώς μπορούμε να έχουμε τις τεχνικές δυνατότητες και ποια πρέπει να είναι η στοχοθεσία για τις παρακολουθήσεις και φυσικά μας ενδιαφέρει να ξέρουμε ποιος ελέγχει τους ελέγχοντες σε αυτήν την περίπτωση. Ποιος ελέγχει τις μυστικές υπηρεσίες. Κατά πόσο η εθνική ασφάλεια παραμένει μονάχα στεγανή στα πλαίσια των κρατών μελών ή αν πρέπει να υπάρξει και κάποια ευρωπαϊκή αρμοδιότητα για να εξασφαλιστεί ότι αυτές οι κόκκινες γραμμές δεν υπερβαίνονται και τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν για τον τομέα αυτό. Αναφέρθηκε και το θέμα της προστασίας των δεδομένων και αναρωτιέμαι αν τα κράτη-μέλη μέσα σε, στα πλαίσια διμερών συμφωνιών μπορούν να έχουν ε, ουσιαστικά παράκαμψη των ε, συμφωνιών για την προστασία των δεδομένων και μέσω διμερών συμφωνιών μυστικών υπηρεσιών μπορούν να τα παρακάμπτουν όλα αυτά. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα δεδομένα τα οποία είναι τα πιο ευαίσθητα και φυσικά μας ενδιαφέρει και στα πλαίσια της προστασίας των δεδομένων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ Μπριγκίτα. Το τελευταίο αυτό σημείο που θέλει να κάνει ο Γιάνν Άλμπερτ και θα σας ζητήσω να κάνετε την τελική σας ε, απάντηση σε όλα αυτά ο Γιάννα Άλμπρεχτ. Απλώς και μόνο για να επανέλθω σε αυτά που είπε η κυρία Ζίπελ. Θα ήθελα να ξέρω αν έχετε κάποιες ε, γνώσεις σε σχέση με συμφωνίες αυτού του είδους που έχουν να κάνουν με τα προγράμματα όπως το PRISM και το TEMPORA σε σχέση με αυτή τη μαζική παρακολούθηση που μας ενδιαφέρει εδώ. Δεύτερον, Μιλάμε και για επιθέσεις στον κυβερνόχωρο. Το GCHQ έχει κάνει επιθέσεις σε συστήματα πληροφορικά αμερικανικών εταιριών, αλλά όπως ξέρουμε και στην Belgacom έχει γίνει κάτι αντίστοιχο στα συστήματα της Belgacom και στους παρόχους υπηρεσιών της Belgacom. Όταν πρόκειται λοιπόν για νομοθεσία κυβερνοεγκλήματος, θα ήθελα να ξέρω κατά πόσο υπάρχει παραβίαση αυτής της νομοθεσίας στα κράτη-μέλη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς παραβιάζεται και η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το κυβέρνο έγκλημα και όταν πρόκειται για τα δικά μας συστήματα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί και εμείς χρησιμοποιούμε τα συστήματα της ΣΥΣΚΟ όλοι μας. Είναι προφανές ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος τα στοιχεία αυτά που των επικοινωνιών μας να έχουν διαβρωθεί. Ποιες είναι οι δυνατότητες λοιπόν εμείς να ζητήσουμε θεραπεία στα δικαστήρια λόγω αυτών των παραβιάσεων των ε, δικαιωμάτων μας και των προσωπικών μας δεδομένων. Αν πρόκειται και για μια παραβίαση των συνθήκων, θα ήθελα να ξέρω ποιες νομικές δυνατότητες έχουμε. Ευχαριστώ. Είναι ενδιαφέρον που λέτε ότι το ερώτημα σας είναι ενδιαφέρον. είδατε, την έρευνά μας για την Belgacom. Βέβαια εγώ δεν τα έχω κοιτάξει, δεν ξέρω αν το είδατε, αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις. Μήπως θέλετε να βγάλετε κανένα συμπέρασμα και ο ένας και ο άλλος. Ευχαριστώ πολύ. Τρία συμπεράσματα. ή μάλλον τρία ερωτήματα. Πρώτα για τις τηλεπικοινωνίες. Έχουμε στοιχεία ότι οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών έχουν γίνει στόχος της GCHQ και άλλων κατασκοπευτικών υπηρεσιών. Είναι λοιπόν πολύ πιθανόν αν μια εταιρεία δώσει στοιχεία σε μια κατασκοπευτική εταιρεία να έχει δώσει και σε άλλες. Ισχύει και για, τον Belgacom και, για την Belgacom και για άλλες τηλεπικοινωνιακές εταιρείες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα, οι τεχνικές μορφές αντίστασης. Εγώ δεν είμαι τεχνικός, αλλά η λύση που διαβλέπουμε όταν συζητάμε με πυρογνώμονε είναι να χρησιμοποιείται λογισμικό open source Uh, uh, γιατί εκεί γίνονται όλα εθελοντικά η ανάπτυξη του λογισμικού δηλαδή και βασικά η υποκλοπή αποφεύγεται γιατί ο ίδιος ο κώδικας είναι διαθέσιμος και οποιοδήποτε έχει τις γνώσεις μπορεί να τον εξετάσει και να δει αν υπάρχουν ε, ευαίσθητα ή αδύνατα σημεία. Αυτό λοιπόν πρέπει να είναι το λογισμικό που πρέπει να ενθαρρύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο. Και αυτό μπορεί ίσως να λύνει και μερικά από τα προβλήματα των επικοινωνιών. Και τώρα για το ερώτημά σας για τη μαζική επιτήρηση και τις απειλές που μπορεί αυτή να επιφέρει. Τα γεγονότα της 11 ης Σεπτεμβρίου ε, έδωσαν την ευκαιρία στους εθνικούς προϋπολογισμούς να χρησιμοποιήσουν πολύ περισσότερα χρήματα για κατασκοπία. Δεν άρχισε αμέσως βέβαια μετά την 11η Σεπτεμβρίου αυτή η δραστηριότητα, αλλά Λίγο πολύ τα τελευταία 3-5 χρόνια έγινε αυτή η έκρηξη και οι αποκαλύψεις δείχνουν ότι το DCHQ e έχει παίξει ουσιώδη ρόλο για την υποβοήθηση κατασκοπευτικών υπηρεσιών και για την παράκαμψη της νομοθεσίας. και ίσως εδώ μάλλον σε κοινωνιολογικό επίπεδο ένας από τους συντάκτες μελέτης ο Μπίγκο δείχνει ότι η συλλογή τεραστίων ποσοτήτων πληροφοριών είναι μια από τις δικαιολογίες που χρησιμοποιούνται για τις καπασουπαευτικές υπηρεσίες για να συνεργαστούν με τους προμηθευτάς. Αλλά ένας άλλος λόγος είναι να μπορούν οι πληροφορίες να ανταλλάσσονται και με άλλες υπηρεσίες και άρα βλέπουμε έναν ανταγωνισμό για όλο και περισσότερη, μεγαλύτερη συλλογή πληροφοριών για να μπορεί κάθε υπηρεσία να θεωρείται ανταγωνιστική της άλλης. Και βέβαια αυτό ζημιώνει τον Ευρωπαίο πολίτη. Σταματάω εδώ και ας μιλήσει ο Σέργιος. Ένα από τα στοιχεία που φάνηκαν από τη συζήτηση είναι ότι εδώ μιλάμε για ενωσιακές αξίες, ένομη τάξη κλπ. Η αντιπρόεδρος Ρέντινγκ είχε μελετήσει το θέμα του άρθρου 7 της συνθήκης και διαπιστώνουμε ότι υπάρχει συστηματική παράκαμψη και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ορισμένες χώρες μέλη. Το θέμα είναι πολύ δύσκολο νομικά γιατί έχουμε πολύ κατακαιρματισμένο νομικό κλίμα. Και βλέπουμε από τη μελέτη ότι μερικές φορές μπορεί αυτό να έχει εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των κατασκοπευτικών υπηρεσιών. για να παρακάμψουν την ισχύουσα νομοθεσία. Αυτό θα έπρεπε να μας ανησυχεί. Για το προηγούμενο δε ερώτημα, επίσης στη μελέτη ζητάμε μόνιμη εφαρμογή μιας υποδομής στην Ένωση που να διασφαλίζει την παρακολούθηση αυτών των αποκαλύψεων για να υπάρχει μια πιο βιώσιμη επιτήρηση και λογοδοσία όχι μόνο όσων γνωρίζουμε τώρα αλλά και των στοιχείων που μπορεί να γνωρίσουμε τους επόμενους μήνες. Και αυτή η υπηρεσία ή η υποδομη θα μπορούσε να συζητήσει και τρόπους αντίδρασης. Αναφέρθηκε το θέμα των εποπτικών αρχών σε εθνικό επίπεδο καθώς και των χειριστών των στοιχείων και cloud computing. Αλλά για τι πληροφορίες μιλάμε, τι στοιχεία. Και εδώ πρέπει να βρεθεί κάποια μεγαλύτερη νομική σαφήνεια. Οι διοκτικές αρχές, το αναφέρει και αυτό η μελέτη, δεν είναι σαφές ποιες είναι. Και αυτό βέβαια υπονομεύει τον βαθμό ευθύνης και λογοδοσίας και κάτι άλλο που φάνηκε από προηγούμενες μελέτες μας είναι ότι ίσως θα έπρεπε να υπάρχει μία μόνιμη επιτροπή για εσωτερικά θέματα που να συζητάει και το θέμα της επιτήρησης της Ευρωπόλ και άλλων παραγόνδων που ασχολούνται με τέτοια θέματα. Και εδώ το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πολύ Σέρτζο. Πολύ Ε, γνωρίζουμε ε, το έργο σου και το εκτιμούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και τους δύο και τον κύριο Ρακάτζη. Ε, είχατε πάρα πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή σας για να εκπονήσετε αυτή τη μελέτη και πραγματικά είναι πολύ χρήσιμο για μας. Και τώρα θα μας βοηθήσει πολύ στην εργασία για την εκπόνηση της δικής μας έκθεσης. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η συνάντηση που είχαμε μαζί σας για ανταλλαγή απόψεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα να πω στους συναδέλφους ότι η επόμενη συνεδρίαση, μάλλον οι ψηφοφορίες σε λίγο θα αρχίσουν στις 12 και 4, δεν θα προεδρεύσω εγώ, θα με σώσει κάποιος αντιπρόεδρος. Ή ο πρόεδρος. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Δυστυχώ είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε αυτές τις συνεδριές πέμπτη και μάλιστα και πέμπτη απόγευμα. Ε, δεν είναι το πιο εύκολο, αλλά για λόγους χρονοδιαγράμματος έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, σα ευχαριστώ και πάλι που ήρθατε και χαίρετε. Uh, um, Α, συγγνώμη, ε, έχω και άλλη ανακοίνωση. Ψηφίζουμε στις 12 και 4, το ξέρετε. Κάποιο αντιπρόεδρο θα έρθει να με σώσει, είπα. Δεν θα προεδρεύσω εγώ. Αλλιώς θα αναγκαστώ να προεδρεύσω και στις ψηφοφορίες. Ε, τι να κάνω, θα το καταπιώ και αυτό. Και αν με θέλετε και τίποτα άλλο, είμαι στη διάθεσή σας. <laughs>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

Good afternoon. Γεια σας. Θα ξεκινήσουμε την ψηφοφορία μας. Έχουμε δύο θέματα που πρέπει να ψηφίσουμε. Το πρόγραμμα για τα δικαιώματα των πολιτών που είναι θέμα της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και έχουμε το κοινό πρόγραμμα με την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων που είναι το νομικό πρόγραμμα. Για το πρώτο θέμα λοιπόν, για το δεύτερο βέβαια θα υπάρξει κοινή ψηφοφορία και από τα μέλη της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων που είναι παρόντα. Ελπίζω ότι έχουμε απατία. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με το πρόγραμμα για τα δικαιώματα των πολιτών. Όπως βλέπετε στον κατάλογο, έχουμε το κείμενο συμβιβασμού. Και αν δεν υπάρξει υποστήριξη του κειμένου συμβιβασμού, θα πρέπει να συνεχίσουμε λεπτομεριακή ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ λοιπόν του κειμένου συμβιβασμού. Θέλω εδώ χέρια. Κατά αποχές. Έχουμε λοιπόν υποστήριξη του κειμένου συμβιβασμού και τώρα η τελική ψηφοφορία με ηλεκτρονική ψηφοφορία. And vote electronically. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο του κειμένου όπως έχει τροποποιηθεί. Άρχεται η ψηφοφορία. Ο κύριος Μπελίνγκουερ δεν έχει κάρτα. Ναι αλλά είναι υπέρ και αυτός. Ωραία. Σας ευχαριστώ. 25 υπέρ, 2 κατά και καμία αποχή. Και θέλω να ευχαριστήσω σε όλους οι οποίοι συνέβαλαν στο θέμα αυτό, στους χειώδεις εισηγητές και στους εκπροσώπους των διαφόρων γνωμοδοτικών επιτροπών για το θέμα αυτό. Και τη Μαρία βέβαια. Και τη Μαρία. Η οποία εργάστηκε πολύ σκληρά για το θέμα αυτό. Μπράβο Μαρία. Σας ευχαριστώ. Και τώρα θα πάμε στο επόμενο θέμα που είναι το κοινό πρόγραμμα για, τα, για το πρόγραμμα δικαστικού χαρακτήρα. Ψηφίζουμε λοιπόν καταρχήν το κείμενο συμβιβασμού. Θέλω να καλωσορίσω όλους αυτούς που είναι παρόντες εδώ. Μήπως θέλετε να πείτε κάτι. Όχι. Υπέρ του κειμένου συμβιβασμού. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν το κείμενο αυτό. Και τώρα ηλεκτρονική ψηφοφορία για το κείμενο όπως έχει τροποποιηθεί, ηλεκτρονικά όμως. Ηλεκτρονικά. Ωραία. 27 υπέρ, μία ψήφο κατά, καμία αποχή. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για την ψηφοφορία. Θέλετε να πείτε κάτι κύριε Μπελίγκουερ. Όχι, τίποτα. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστώ πολύ.